Καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες. Ξεκινάμε νωρίτερα από τη συνήθως, 14 ε, και 30, για πολλούς λόγους. Αποτελεσματικότητα το ονομάζουμε. Εδώ παρακαλώ να είστε έτοιμοι με την κάρτα σας και να δείτε αν λειτουργούν τα μηχανήματα για να περάσουμε απευθείας στην ψηφοφορία και να ψηφίσουμε πρώτα τη γνωμοδότηση για την ε, ε, Air France κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση επί τα απέτηση της Γαλλίας. Είναι ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται αυτή, πέρας. 29 προς μία ψήφο. Δεύτερον, κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής. Άρχεται η ψηφοφορία για τη δεύτερη υποστολή αυτή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, Πέρα αυτή. 32 προς 1. ερώτημα με αίτημα προφορική απάντηση σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την επισφαλή απασχόληση. Τα ζητήσαμε και με τους συντονιστέ Υπέρ. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. να κάνουμε έλεγχο για την δεύτερη τροπολογία. Έρχεται αυτή. Πέρας για την τροπολογία 2. 21 ψήφοι υπέρ, 16 κατά. Τελική ψηφοφορία για την ερώτηση με έτοιμα προφορικής απάντησης, όπως τροποποιήθηκε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 37 ψήφους ε, υπέρ, καμία κατά. Και τώρα έκθεση Μπέκερ. Καταστατικό επιχειρήσεων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Ε, συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 να κάνουμε έλεγχο ηλεκτρονική ψηφοφορία έρχεται πέρας 37 εγκρίνεται με 22 προς 18 ψήφους. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 56 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 14, συμβεστική 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 99 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 συμβαστική 17 υπέρ κατά Δεν είδα αρκετά χέρια. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 109. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική όχι. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ετεολογικές σκέψεις, συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 3 Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, 20, 20, με συγχωρείτε, 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, να ελέγξουμε την 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Και μετά ψηφίζουμε για το σχέδιο γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 40 υπέρ, 3 κατά. Να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε στην ακρόαση. Σαφείς και προβλέψιμες εργασιακέ συνθήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς να καλωσορίσω θερμά όλους τους ε, προσκεκλημένους μας τους εμπειρογνώμονές μας που υποδεχόμαστε, οι οποίοι θα μοιραστούν μαζί μας τις δικές τους ε, γνώσεις και εμπειρίες. Δυστυχώς, η κυρία Καλβέτσα Τσαμπών, μάλλον συγγνώμη, ο κύριος Μπένιο δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα. και η κυρία Κάσα Μπαμόντε. Ε, υπήρξαν κάποιε απεργίε στι αερογραμμέ, όχι ο κύριο Καλβετσαμπών. Ε, στα τέλη τη περασμένη χρονιά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή τη για διαφανή σαφείς και προβλέψιμε εργασιακές συνθήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόταση η οποία ασχολείται με δύο συνιστώσεις, την αξιολόγηση της σχετικής οδηγίας και τις δημόσιες διαβουλεύσεις για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, που υπογραμμίζει την απόσταση μεταξύ του ισχύοντος κοινωνικού κεκτημένου και των προσφατότερων εξελίξεων στην αγορά εργασίας. Αυτό τονίστηκε και στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου τον Ιανουάριο του 2017 για τον κοινωνικό πυλώνα και πέραν του ψηφίσματος του, του Ιλίου 2017 για τις εργασιακές συνθήκες και την επισφαλή εργασία, το Κοινοβούλιο απίθυνε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, αναθεωρήσει την οδηγία για να λάβει υπόψη στην παράτυπη εργασία. Η Η ε, οδηγία για τι ε, ελάχιστε δηλώσει θα πρέπει να προβλέπει τουλάχιστον ένα ελάχιστο εργασιακών συνθήκων, ένα ελάχιστο εργασιακών δικαιωμάτων και βάσει τη ε, νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημερινή ακρόαση έχει σκοπό να συνεισφέρει στην μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόταση αυτή και όπως όλοι γνωρίζουμε σε αυτή την Επιτροπή είναι μεγάλη σημασία για την κοινή γνώμη Έχουμε τον εισηγητή, τον κύριο Καλβέτ τα μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης, που έχουν προετοιμαστεί για αυτήν την συζήτηση προκειμένου να δούμε τι ενδιαφέρει τους βασικούς, τι απασχολεί τους βασικούς ενδιαφερομένους εδώ. Θα ήθελα να παρουσιάσω τον πρώτο μας ομιλητή, τον κύριο Ρόλφ Κλάισνερ, Διευθυντή για την Κοινωνική και Πολιτική και Πολιτική Υγείας για το Ευρωπαϊκό Ομοσπονδιακό Εμπορικό Επιμελητήριο, Οικονομικό Επιμελητήριο και σας παρακαλώ να πάρετε το λόγο για την παρουσίασή σας. Thank you very much for... Ευχαριστώ πολύ που μου κάνετε αυτή την τιμή να σας παρουσιάσω την κατάσταση όσον αφορά την αυστριακή οικονομία τα έχω στα αγγλικά εδώ γραμμένα, αλλά θα σας τα πω στα γερμανικά. Λοιπόν, ξεκινάμε με την πρόταση της οδηγίας. Καταρχήν η οδηγία διαφοροποιείται σημαντικά από την ε, οδηγεί απόδειξης ε, που πρέπει να αντικαταστήσει και ξεκινάει με το πεδίο εφαρμογής όπου υπήρχαν εξαιρέσεις ε, που τώρα διαγράφονται ε, και τώρα αναφέρονται περιπτώσεις πολλών εποχικών θέσεων εργασίας και μικρής διάρκειας. Αυτές όλες καλύπτονται. Θεωρούμε λοιπόν ότι όλη αυτή η προσπάθεια είναι τεράστια σε σχέση με το αντικείμενο. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι οι σχέσεις απασχόλησης που δεν υπερβαίνουν σε διάρκεια τον ένα μήνα πρέπει να εξαιρούνται. Περνάω λοιπόν τώρα σε ένα σημαντικό θέμα που αφορά στον ορισμό της έννοιας εργαζόμενος. Η πρόταση που έχει κατατεθεί ανάγεται σε κάποια παραδείγματα. Διότι καταρχήν γίνεται ορισμός του εργαζόμενου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέχρι τώρα οι οδηγίες ε, αφορούσαν εθνικούς ορισμούς. Ε, στην νομολογία όμως ε, δεν υπάρχει κανένας σημαντικότερος διαχωρισμός ανάμεσα στους μισθωτούς και τους επιτιδευματίες όχι μόνο στο εργατικό και το φορολογικό δίκαιο, αλλά και σε άλλους τομείς. Προκύπτει εξή εξήγηση. Η προάγονται όλο και περισσότερο θέσει απασχόλησης μη επισφαλής. Αν δούμε όμω ε, κάποιες μελέτες και αυτήν του Eurofond, πρέπει να πούμε ότι υποχωρούν ή ε, παρουσιάζεται στασιμότητα στι μη τυποποιημένες θέσει απασχόλησης. Και γι' αυτό επειδή έχουμε αυτή τη βάση, κάναμε και το επόμενο βήμα. Και ανακαλούμε ή βασιζόμεθα σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που κατά την άποψή μας οι αποφάσεις αυτές είναι αρκετά απαρχιωμένες. Η μία αφορά την ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων και η άλλη αφορά ε, το, την, το άτομο, την οντότητα που ισούται με εργαζόμενο. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό μπορεί να χρησιμεύσει ως ορισμός του εργαζομένου. Όσον αφορά τη δική μου τη χώρα, ο ορισμός αυτός, αυτή η πρόταση είναι ευρύτερη από αυτό που κατανοούμε εμείς στην Αυστρία ως εργαζόμενο. Για μας παίζει ρόλο η οικονομική ε, εξάρτηση ε, και ρόλο παίζουν ε, ο τρόπος εργασίας, ε, η μορφή της απασχόλησης. Όλα αυτά εντάσσονται μέσα στον ορισμό της έννοιας επιχείρηση. Στην Αυστρία η έννοια εργαζόμενος δεν περιλαμβάνει τους freelancers και παρεμφερείς εργαζόμενους. Αυτό το παρεμφερείς στην Αυστρία ταυτίζεται σχεδόν με τον ορισμό του εργαζόμενου σε, αυτή την οδηγία. Ε, παρεμφερείς απασχολούμενοι στην Αυστρία δεν τους αφορά αυτή η οδηγία και αυτό είναι με σημαντική παρέμβαση, τουλάχιστον στην Αυστρία. Γιατί άτομα που δεν είναι εργαζόμενοι, για αυτούς δεν ισχύει το εργατικό δίκαιο ε, και κυρίως δεν ισχύει το ωράριο εργασίας. Όμως με την οδηγία θέλουμε να ρυθμίσουμε το ωράριο εργασίας. Θα ήθελα να σε επισημάνω και κάποια άλλα προβλήματα που ανακύπτουν. Δηλαδή στο μέλλον θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για τις ε, προϋποθέσεις καταγγελίας της σύμβασης, οι οποίες ε, προϋποθέσεις είναι αρκετά περίπλοκες ε, και προκύπτουν από διάφορους κανονισμούς, παραδείγματος χάρη για άτομα με αναπηρία, για πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους, προκύπτει μια ισότητα και γι' αυτό όλο αυτό είναι περίπλοκο. Εξάλλου, όσον αφορά τους, το χρόνο εργασίας πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα σχέδιο που είναι γνωστό μόνο στην Αυστρία ε, και όχι σε άλλες χώρες γιατί στην Αυστρία υπάρχουν και συμβάσεις μηδενικής απασχόλησης, μηδενικού, μηδενικών ορών και θα επανέλθω να σε εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Αυτά λοιπόν πρέπει να δοθούν ως πληροφορίες την πρώτη μέρα. Παλαιότερα μπορούσε να γίνει και αργότερα. Όμως στην πράξη πριν ξεκινήσει κανείς να εργάζεται ε, πρέπει να συμφωνήσει με τον εργοδότη για τα σημαντικότερα θέματα, ας πούμε για το ωράριο ή για τις απολαβές. Πολλές φορές όμως ε, τέτοιου είδους ε, θέματα διευκρινίζονται και κατά την πρώτη εβδομάδα της εργασίας που σε τελική ανάλυση οι πληροφορίες αυτές δίδονται αρκετά καθυστερημένα, γι' αυτό για μας είναι σημαντικό να υπάρχει ένα περιθώριο ενός μηνός για να μπορεί και να ε, το πράττει ο εργοδότης να ενημερώνει τον εργαζόμενο. Περνάω στο άρθρο 8 απασχόληση πολλών μορφών. Εδώ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του κανείς ότι ο εργοδότης είναι υπεύθυνο για το ωράριο εργασίας και ο εργαζόμενος, αν έχει εργαστεί και σε άλλη απασχόληση, αυτό θα πρέπει να το γνωρίζει ο εργοδότης και να περιορίζει το ωράριο εργασίας ή την απασχόληση του εργαζόμενου σε κάποιον άλλο τομέα. Πάω τώρα στο άρθρο 9 που ρυθμίζει το ωράριο εργασίας και αυτό το άρθρο 9 έμεσα αφορά τις συμβάσεις μηδενικών ωρών που ανέφερα και προηγουμένως. Και εδώ προκύπτουν σημαντικές συνέπειες αν δεν αναφέρονται οι ώρες εργασίας. Και στην Αυστρία τουλάχιστον αυτό περιορίζει την ευελιξία. Γιατί, Γιατί στην Αυστρία είναι δυνατόν να επιβάλλονται υπερορίες και εκτός του κανονικού οραρίου. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν, αν δεν υπάρχει καταμέτρηση των κανονικών ωρών εργασίας, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν και περιορίες. Και αυτό ε, θα περιορίζει την ευελιξία. Εγώ παραδείγματο χάρη θα γυρίσω σπίτι μου μάλλον το βράδυ, που είναι εκτός ωραρίου εργασίας μου. Ε, θα μπορούσα να έχω αρνητή να έρθω εδώ, γιατί στη σύμβαση εργασίας μου ε, δεν αναφέρει ότι θα πρέπει να δουλεύω και να εργάζομαι και το απόγευμα ή το βράδυ. Κατά τα άλλα, το άρθρο 9 αφορά σε άτομα τα οποία μπορούν να εξαιρούνται από την οδηγία περιεργασίας, δηλαδή ε, τους οικείους του εργαζόμενου και τα στελέχη της εταιρείας. Άρθρο 10. Κατά την άποψή μας αυτό δημιουργεί προβλήματα διότι η έννοια ε, προβλέψιμος και περισσότερο ασφαλής ε, αυτά τα επίθετα δεν προσφέρουν εγγύησης και μπορεί οι επιχειρήσεις πολύ συχνά να εξαναγκαστούν να τοποθετηθούν και να ενημερώσουν. Προχωρώ πιο κάτω Περνάμε στο άρθρο 11. Για μένα εδώ ε, υπάρχει κάποια σάφια. Πρόκειται για την εκπαίδευση και για την υποχρέωση της δωρεάν εκπαίδευσης. Και τίθε το εξή ερώτημα. Ο εργαζόμενος δεν καταβάλει το αντίτιμο των κύκλων μαθημάτων ή το καταβάλει και μετά το δικαιούται στην Αυστρία ε, ήθιστε ο εργοδότης ε, να πληρώνει για την εκπαίδευση του εργαζόμενου. Αν όμως ε, καταγγελθεί νωρίτερα η σύμβαση, τότε ο εργαζόμενος πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα της εκπαίδευσης, γιατί ο εργοδότης δεν ωφελήθηκε από την εκπαίδευση, αλλά ωφελήθηκε ο ανταγωνιστής του. Και για μένα εδώ υπάρχει κάποια σάφια και πρέπει να διευκρινιστεί. Πάω τώρα σε ένα άλλο σημαντικό σημείο, διότι στην Αυστρία υπάρχουν σε όλη την Αυστριακή επικράτεια συλλογικές συμβάσεις για όλους τους εργαζόμενους. Το άρθρο 12 επιτρέπει αποκλήσεις από συλλογικές συμβάσεις και εδώ είναι πολύ σημαντικό να μην γίνεται αναφορά σε νέες συλλογικές συμβάσεις, αλλά σε ήδη υπάρχουσες συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες προβλέπουν ε, τα θέματα δικαιώματα του ωραρίου εργασίας και πάρα πολλά συναφή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί στην Αυστρία υπάρχουν συμβάσει, σε τι οποίε διαπραγματεύονται αν θέλετε τα συνδικάτα με τα οικονομικά επιμελητήρια. Περνάμε τώρα στο άρθρο 13 το οποίο άρθρο αναφέρει όλα τα επίπεδα στα οποία ρυθμίζεται το εργατικό δίκαιο όλα αυτά οφείλουν να εφαρμόσουν την οδηγία. Κατά την άποψή μου αυτό δημιουργεί προβλήματα, κυρίως διότι η οδηγία ή αν θέλετε η πρόταση πρέπει να ισχύει ήδη για ε, υπάρχουσες ε, συμβάσεις και όχι για μελλοντικές συμβάσεις ή νέες συλλογικές συμβάσεις. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι εδώ γίνεται παρέμβαση στην αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και παρέμβαση σε ήδη υπάρχουσες συμβάσεις επανέλθω αυτό. Άρθρο 14. Το άρθρο αυτό ε, συνεπάγεται νέα εργαλεία, νέα παραδείγματα, για να το πω έτσι απλά, ε, προβλέπεται η αντιστροφή του βάρους απόδειξης και αυτό μπορεί να είναι πολύ σοβαρό. Αν μια επιχείρηση ε, δεν δώσει μία πληροφορία για οποιοδήποτε λόγο, ε, παραδείγματο χάρη ε, να μην γνωρίζει ο εργαζόμενος ε, κατά πόσον μία σύμβαση είναι χωρίς χρονικό περισμό, Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Θα πρέπει λοιπόν να επιβληθεί στα κράτη-μέλη να λαμβάνουν μέτρα έτσι ώστε να εφαρμοστεί η οδηγία. Σε τελική ανάλυση όμως τα μεμονωμένα εργαλεία, το πώς ακριβώς θα γίνεται αυτό στην πράξη, ε, αυτό να εναπόκειται στα κράτη-μέλη και να μην είναι απαραίτητο να ισχύει η αντιστροφή του βάρους απόδειξης ή να είναι απαραίτητο να επιβάλλονται πρόστιμα. Στην Αυστρία υπάρχουν ε, ε, συλλογικές συμβάσεις όλη την επικράτεια. Όλοι οι εργαζόμενοι εντάσσονται στον ε, ένα είδους εργατικού συλλόγου και έτσι έχουν δικαίωμα σε συγκεκριμένα δικαιώματα. Τελειώνω σιγά σιγά, πάω στο άρθρο 17, το οποίο άρθρο 17 ρυθμίζει την προστασία από καταγγελία σύμβασης. Κατά την άποψή μου αυτό χρειάζεται μια διαφορετική βάση, ε, χρειάζεται την ομοφωνία διότι βεβαίως ε, οι κανονισμοί για καταγγελία σύμβασης είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι. Οι κανονισμοί αυτοί αφορούν όχι μόνο εργοδότη εργαζόμενο, αλλά αφορούν και την αγορά εργασίας. Παράδειγμα, το άρθρο 17 προβλέπει ότι ορισμένες ε, άδικες καταγγελίες πρέπει να απαγορεύονται, αλλά στην Αυστρία ήθιστε ως εργαζόμενος ε, να έχει κανείς το δικαίωμα να προσβάλλει τις καταγγελίες αλλά έχει ε, διαφορά το κατά πόσο αυτό επιτρέπεται ή απαγορεύεται. Πάντως ε, μπορούν να προσβληθούν ε, οι συμβάσεις στο δικαστήριο. Στην Αυστρία δεν ισχύει αυτή η νοοτροπία hire and fire και αυτό είναι ένας λόγος που σε εμά λειτουργεί εύρυθμα η αγορά εργασίας. Ε, το άρθρο 21 αυτό πρέπει να ισχύει και για ήδη υπάρχουσες ε, συμβάσεις. Εμείς όμως αυτό το βρίσκουμε προβληματικό γιατί στην Αυστρία εμείς έχουμε βελτιώσει κάποιες ρήτρες συμβάσεις αλλά αυτό το κάναμε για νέες συμβάσεις και λέμε οι εργαζόμενοι οι οποίοι καλύπτονται από παλαιές ε, συμβάσεις αυτοί κατά κανόνα είναι πολύ καλά προστατευμένοι και είναι άδικο αν πρέπει κανείς να παρέμβει στο κείμενο δίκαιο. Ε, αν χρειάζεται παρέμβαση, τότε κατά κανόνα σε νέες ε, συμβάσεις. Περνάω τώρα στο συμπέρασμά μου. Η πρόταση που έχει κατατεθεί περιλαμβάνει ε, κτεταμένα ε, δικαιώματα και διατάξεις εφαρμογής που αλλάζουν την μέχρι τώρα οδηγία η πρώτη περιλαμβάνει νέα παραδείγματα, αποτελεί ουσιαστική παρέμβαση στο εθνικό δίκαιο. Για άλλη μια φορά, ο ορισμός του εργαζόμενου, τα όρια ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτό είναι το σημαντικότερο όριο που υπάρχει στην νομολογία και νομίζω ότι ε, θα πράξουν πάρα πολλά προβλήματα εάν τελικά προκύψει σύγκρουση των ορισμών των εθνικών με των ενωσιακών. Κατά τη δική μας λοιπόν άποψη αυτή η πρόταση δεν συμβαδίζει με τους στόχους του REFIT, που είναι να περιοριστεί η γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις, ε, κυρίως για τις μικρές επιχειρήσεις, που είναι και οι περισσότερες του δικού μας του οικονομικού επιμελητηρίου. Στόχος επίσης είναι η αύξηση της διαφάνειας που ούτε και αυτός επιτυγχάνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ, λέει Πρόεδρος. Τελειώσατε, τελειώσατε. Πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μα ε, είπατε για το να δώσουμε τον ε, λόγο στον κύριο Νίλ Στραμπ που είναι ο πρόεδρος ε, του Chair, που είναι πρόεδρο μάλλον τη Business europe Industrial Relations, δηλαδή των εργασιακών σχέσεων Business Europe. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι περίπλοκη αυτή η οδηγία. Οπότε χρειάζεται κανείς όσο μπορεί παραπάνω. Και η εντύπωση μας είναι ότι αυτό αφορά κάποιους εργαζομένους ε, για τους οποίους υπάρχει ε, ζήτηση και θα επανέλθουμε σε αυτό αλλά τελικά όλοι οι εργαζόμενοι πρόκειται να καλυφθούν και κάποιες διατάξεις, κάποιους με υψηλές δεξιότητες και υψηλή αμοιβή. Οπότε φοβόμαστε ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές και αυτό σημαίνει ότι κάποιες εταιρείες θα είναι λιγότερο πρόθυμες τέτοιους εργαζόμενους να απασχολήσουν ανταυτού θα συνάπτουν συμβάσεις με πλατφόρμες, με παρόχους υπηρεσιών. Δεν πειράζει. Αλλά δεν γίνεται να, να υποχρεώνουμε τι επιχειρήσει να προσλαμβάνουν και από την άλλη μεριά δίνουμε αντικίνητρα. Ο μιλητή μιλά μακριά από το μικρόφωνο το οποίο το έχει γυρίσει σε άλλη κατεύθυνση και δεν ακούγεται καλά. Οπότε, τώρα έχουμε αυτούς οι οποίοι εμείς δεν, δεν ε, ε, ε εκπροσωπούμε εργαζομένους, αλλά ε, εταιρείε, εργοδότες Οπότε κάποιο τρόπο πολλές φορές έχουμε να λύσουμε συγκρούσεις και ανταγωνισμό μεταξύ διαφόρων μορφών απασχόλησης. Οπότε και αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, είναι να υπάρχουν θεμητοί όροι ανταγωνισμού ε, στον χώρο αυτό. Κατά δεύτερο λόγο, συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, ξεκάθαρη σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου όσον αφορά δικαιώματα και υποχρεώσεις για αυτήν την εργασιακή σχέση. Και για αυτό τον λόγο και εμεί. Από το 1991 και μετά ήμασταν ε, ε, υπέρ αυτής της οδηγίας προς για την υποναθεώρηση και συμφωνούμε με την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρούμε ότι συνεχίζει και αποδίδει αυτή η νομοθεσία. Αυτά αν τα λάβετε υπόψη επίσης τώρα χρειάζεται να εξυγχρονίσουμε αυτή την οδηγία του 1991 για να έχουμε έτσι μια ε, ιστορική άποψη. Πάντως πριν ε, σας πω τις απόψεις μας για την ε, πρόταση της Επιτροπής, ίσως ε, θα πρέπει να δούμε γιατί οι κοινωνικοί εταίροι δεν έκαναν διαπραγματεύσεις μαζί μας. Μα γιατί για το refit χρειάστηκαν δύο χρόνια. Μετά πέρασε άλλος ένας χρόνος μέχρι να διαβουλευτούμε έξι εβδομάδες μετά την αρχή των διαβουλεύσεων ζητήσαμε για διερευνητικές συνομιλίες και μας είπε η Επιτροπή ότι δεν συμφωνεί με αυτό και ότι πρόκειται να κατεβάσει την πρότασή της μέχρι τα τέλη του έτους. Οπότε μας, μας τρίμωχνε. Δηλαδή θέλαμε να διαπραγματευτούμε, αλλά δεν μας δόθηκε ευκαιρία να το πράξουμε γιατί υπήρχε αυτή η πίεση χρόνου. Τώρα δεν μπορώ να τα καλύψω όλα στα 10 λεπτά που μου δώσατε. Ε, άλλωστε ο κύριος ε, Γκλάισνερ ε, είπε πολλά. Επομένως δεν θα σας πω για τον ευρωπαϊκό ορισμό του εργαζομένου, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για τι θα πρέπει να κάνουν οι πολιτικοί, τι πρέπει να κάνουν οι κοινωνικοί εταίροι, γιατί συνεχώς μεταβάλλεται η αγορά απασχόλησης. Κανείς μας δεν μπορεί να προβλέψει σε 5-10 χρόνια τι μορφή θα έχουν οι εργασιακές σχέσεις. Άρα θα πρέπει όλοι να προβούν σε κάποιο είδους ε, επανασχεδιασμό του τι θα πει εργοδότη, του ορισμού δηλαδή εργοδότη και εργαζομένου. Έχουμε και τον έμεσο εργοδότη επίσης και δεν καταλαβαίνουμε ούτε συμφωνούμε με την σχετική πρόταση γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι θα πρέπει ο εργαζόμενος να ξέρει ποιος είναι ο εργοδότης του. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές πιθανότητες αλλά μόνο μία. Άρα δεν συμφωνούμε με την πρόταση της Κομισιόν επ' αυτού επίσης. Εάν υπάρχουν κάποιες ε, επιφυλάξεις για το τι γίνεται με τα κράτη-μέλη και συμφωνούμε με αυτά που λέει η Κομισιόν, τα κράτη-μέλη θα πρέπει, αν υπάρχουν επιφυλάξεις, να μπορούν να ξεχωρίσουν το ποιος είναι ο εργοδότης. Να μην υπάρχει επομένως η έννοια του έμεσου εργοδότη. Τώρα όσον αφορά το ενημερωτικό κομμάτι, μας είπε για την κατάρτιση ο Δόκτωρ Γκλάισνερ. Άρα να προσέχουν υπάρχει εδώ πέρα ε, κάτι παραπλανητικό. Δηλαδή, πολλές φορές η εκπαίδευση είναι κάτι πολύ ευρύτερο του να αποκτά κανείς ε, κάποιους τίτλους, κάποια πιστοποιητικά για την κατάρτισή του. Και ε, είναι θέμα όρων λειτουργίας μιας ε, εταιρεία. και υπάρχει σχετική πολιτική της κάθε εταιρεία και είναι όπως νεοπροσληφθέντες καλύπτονται. Από αυτό επίσης πρότεινε η Επιτροπή θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ αυτών που έχουν προβλέψιμη εργασία και αυτών που δεν έχουν. Αυτό είναι τελείως νέο. Νομικά αυτό δεν προβλέπεται. Ούτε από πώς κάποιος θα χαρακτηρίσει τη δουλειά κάποιου. Να του πει εσύ δουλεύεις ε, προβλέψιμα και ο άλλος όχι. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω πώς να κάνω αυτή τη διάκριση, άρα θα πρέπει εδώ να υπάρχει ασφαλεία δικαίου, να ξέρουμε τι ισχύει στην οδηγία. Τι κάνει κανείς σε μια μέρα εργασία, μια εβδομάδα εργασία και κατόπιν θα πρέπει να διαπιστώνει ακόμα και όταν ε, υπάρχει εργασία εκτός ε, προβλεπομένων ή νομίμων τέλος πάντων ορών απασχόλησης. Αν δεν διορθωθεί αυτό δεν υπάρχει ασφαλή δικαιοτήρα. Τώρα, για τα δικαιώματα. Παράλληλη απασχόληση. Εδώ να σταθούμε γιατί για κάθε εταιρεία θα πρέπει οι σημαντικοί εργαζόμενοι όπως οι μηχανικοί υπολογιστών είναι κάποιοι που η δουλειά τους κοστίζει πολύ στην εταιρεία. Γιατί αν υπάρχει μία βλάβη στους υπολογιστές θα πρέπει να υπάρξει η α, επισκευή που έχουν σημασία αυτές οι εταιρείε θα πρέπει να καλύψουν αυτούς ψηλών δεξιοτήτων εργαζομένων Αυτοί πληρώνονται αδρά από κάποια εταιρεία για να είναι διαθέσιμοι το υπάρξει βλάβη σε επίπεδο ας πούμε πληροφορικής. Τώρα όσον αφορά το επαγγελματικό απόρριτο είπαμε τι ισχύει, θα πρέπει να υπάρχουν αλληλεκτικές όπως προαναφέραμε. Η Επιτροπή εφαρμόζει πάλι αυτή τη διάκριση μεταξύ του τι είναι άκρος προβλέψιμο. Και μιλούμε για αυτούς τους υψηλά που δουλεύουν σε αυτές τις μη προβλέψιμες εργασίες. Πώς να ξέρει κανείς πόσοι δουλειά έχουν. Αν κανείς μας απομακρυνθεί από αυτή την ομάδα, τότε θα δει ότι μιλούμε και θυμίζουμε τη δουλειά αυτών, των υψηλά εμβεβόμενων. Και αυτοί παίρνουν μπόνους, έχουν κάποια ρεπό, αμείβονται για την για την υπερορία τους. Πάντως η Επιτροπή δεν ρυθμίζει ρεαλιστικά εδώ το θέμα. Και είπαμε ότι δεν πρόκειται περί νομικής έννοιας. Άρα πώς θα εφαρμόσει κανείς αυτά που προτείνει η Επιτροπή. Πάλι επομένως πάμε για κενό στην νομοθεσία. Ήδη για την υπάρχουν τρεις οδηγίες, οι οποίες Περιθυμίζω. τα, των διαφορετικών μορφών απασχόλησης, part-time, fixed time κλπ. Υπάρχουν διατάξεις πολύ συγκεκριμένες, ειδικέ για διαφορετικές μορφές εργασίας και προβλέπεται επίσης το πώς γίνεται η μετάβαση από τη μία μορφή εργασίας στην άλλη. Εν προκειμένου όμως είναι γενικό χαρακτήρα η ρυθμίση. Άρα η Επιτροπή θα έπρεπε να λέει ότι αυτά που λέμε εδώ θα πρέπει να ισχύσουν και για τις άλλες μορφές προσχόλησης τα οποία ήδη ρυθμίζουν σε τρεις οδηγίες. Και υπάρχουν επίση και συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων. Άρα με αυτή την πρόταση αναμειγνύεται στη, στάση όσα μας φωνήσει η κοινωνική εταιρεία, αναμειγνύεται σε αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπω και το ρολόι τι θέλετε να κλείσω. Καλά, καλά. Τώρα, όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση κατάρτιση, όποτε είναι υποχρεωτικό να γίνει αυτό για να κάνει κανείς τι αυτή την εκπαίδευση, αυτό αφορά και την ασφάλεια, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο εν προκειμένου. Ότι αφορά υγεία και ασφάλεια. Η εκπαίδευση για υγεία και ασφάλεια αυτή η ρύθμιση, αυτή η διάταξη. Ναι, σωστό είναι αυτό που λέει ότι θα πρέπει να σεβαστεί τη Συμφωνία των Γενικών Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ισχύει ότι έχουν συμφωνήσει διαφορετικό η κοινωνική εταιρεία. Διαφορετικά από την οδηγία όμω δεν καταλαβαίνω γιατί παρεκκλίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τι ε, προηγούμενε οδηγίε. Γιατί περιορίζουν το πεδίο εφαρμογή των συμφωνητών κοινωνικών εταιρών. Συγκεκριμένοι τομεί, συγκεκριμένε περιπτώσει θα μπορούσε να λέει ότι καλύπτει. Όμως τώρα μιλούμε για διατάξεις οριζόντιου χαρακτήρα που ισχύουν για πάσα συλλογική σύμβαση. Ακούσαμε τι ισχύει για την Αυστρία που ισχύει και για άλλες χώρες μέλη. Όλα αυτά επομένως θα πρέπει να τροποποιηθούν. Επίσης, για το άρθρο 13 για τη συμμόρφωση. Α, ήδη ο Δόκτωρ Γκλάσνερ το σχολίασε και η υπόλοιπη οδηγία επίσης σχολιάστηκε από εκείνον. Επίσης να σας πω ότι και θα λες τα δικαιώματα αφορά αυτούς τους υψηλών δεξιότητων και υψηλού αμοιβή. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί εδώ πέρα θα πρέπει να υπάρχει ειδική προστασία όσον αφορά τις απολύσεις. Πώς να τα εξηγήσει αυτά στον ε, κόσμο. Γιατί χρειάζεται ειδική προστασία για τις Εδώ. Αυτά. Ευχαριστώ. Thank Εμείς ευχαριστούμε. Τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Βίπκε Βάρνεκ, νομική σύμβουλο στην ETUC, το Ευρωπαϊκό, ε, την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση δεν αναλύσω άρθρο προς άρθρο την οδηγία, πρότιμο να σταθώ σε ορισμένα σημεία που τα βρίσκω σημαντικά από τη δική μας τη σκοπιά. Πρώτα απ' όλα για την ΕΤΟΚ ε, να πω ότι καλωσορίζουμε την ε, επικαιροποίηση της οδηγίας για τις γραπτές δηλώσεις καθώς και την προφορική αναγγελία ότι η ε, επικαιροποίηση αυτή θα ε, ακολουθήσει τις εξελίξεις των ε, Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Για μας είναι σημαντικό να δούμε ότι με την επικαιροποίηση της οδηγίας αυτής μπορούμε να δώσουμε σάρκα και οστά στα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, στην πράξη. Είμαστε στα χέρια σας λοιπόν, ελπίζουμε αυτό να ολοκληρωθεί πριν τις ερχόμενες ευρωεκλογές, ώστε οι εργαζόμενοι να δουν ότι η οδηγία αυτή θα κάνει κάποια διαφορά στη ζωή τους. Ο στόχος που θέτει η πρόταση της Επιτροπής είναι η προστασία των εργαζομένων. Κατά την άποψή μας χρειάζονται σοβαρές τροποποιήσεις στην οδηγία για να επιτευχθεί σωστά ο στόχος αυτός. Ιδίως για όσους βρίσκονται σε βάλωτη θέση και έχουν επισφαλείς σχέσεις εργασίας. Νίλς, φαντάζομαι ότι ε, καταλαβαίνεις και εσύ, η οδηγία αυτή αφορά περισσότερο εργαζομένους υψηλών προσόντων. Για μας λοιπόν ε, το σχέδιο της ε, οδηγίας δεν επιτυχάνει το στόχο του. Υπάρχουν κενά και υπάρχουν αλλαγές που δεν έχουν γίνει. Οι εργοδότες θα μπορούν να ε, αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους και να μην έχουν την πολυπόθητη προστασία τους οι εργαζόμενοι. Εφόσον ένας εργοδότης έχει βάλει σε ένα χαρτί ε, τις συνθήκε εργασία και τους όρους της σύμβασης και ενημερώσει τον εργαζόμενο, έχει ακολουθήσει αυτά που επιβάλλει η οδηγία. Αλλά πού είναι η προστασία. Εκεί χρειάζεται βοήθεια από το Κοινοβούλιο για να ε, διορθωθεί το κείμενο και να γίνει πραγματικά ένα κείμενο που προσφέρει προστασία. Είμαστε πολύ θετικοί για τη διεύρυνση του πεδίου της οδηγίας. Να περνάμε δηλαδή από τον ε, μισθωτό στον εργαζόμενο, είναι σημαντικό αυτό. Ως προς τον ορισμό, βεβαίως χρειάζεται ορισμός που να προστατεύει επαρκώς ένα τεράστιο ρυθμό ανθρώπων Γνωρίζουμε όλοι ότι σε διαφορετικά κράτη-μέλη προσφέρονται διαφορετικές επιλογές και λύσεις και γι' αυτό πρέπει να φωτογραφίσουμε την κατάσταση αυτή. Υπάρχουν κράτη-μέλη που χρησιμοποιούν κριτήρια και άλλα χρησιμοποιούν εθνικούς ορισμούς. Για μας θα είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι κατεύθυνση θα ακολουθήσετε κι εσείς προς αυτά. Βεβαίως μας δυσκολεύουν οι ε, όροι under the direction, υπό τη διεύθυνση. Θεωρούμε ότι η οδηγία αυτή πρέπει να ε, γίνει, ε, να λάβει υπόψη της και μελλοντικέ εξελίξεις για να αντέξει. Δηλαδή νέες μορφές εργασίας όπως εργαζόμενοι σε πλατφόρμες. Δεν θεωρούμε ότι καλύπτονται από το κείμενο. Και ίσως αντιδρώντας όσοι υπόθηκαν προηγουμένως, για μας οι εξαιρέσεις που ακόμη συμπεριλαμβάνονται, διαφορετικές από το παρελθόν, αλλά και πάλι υπάρχουν εξαιρέσεις, πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά. Αναφερθήκατε στο πακέτο ενημέρωσης και το θέμα του χρονοδιαγράμματος. Για μας βεβαίως πρέπει να προηγηθεί από την εργασιακή σχέση. Και πρέπει να ε, παραδεχτώ ότι προσωπικά δεν καταλαβαίνω πώς σε μια εποχή που όλα γίνονται μέσω μηχανημάτων και διαδικτύου, πώς οι εργοδότες χρειάζονται τέσσερις εβδομάδες για να τα περιλάβουν όλα αυτά σε ένα φύλλο χαρτί. Εάν σκεφτώ τις μικρές επιχειρήσεις τέλος πάντων, ένας εργοδότης δεν προσλαμβάνει κάποιον χωρίς να ξέρει με τι όρος τον προσλαμβάνει. Εμείς ως ΕΤΟΚ ελπίζουμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ε, απαγορευθούν οι συμβάσεις ε, επαναλαμβανόμενες, διότι θεωρούμε ότι οι ευέλικτες και Επισφαλής συμβάσεις δεν πρέπει να είναι ευρωπαϊκό μοντέλο ως προς την προβλεψιμότητα άρθρο 9. Αυτό για μας είναι πολύ ε, σημαντικό, είναι θεμοσίας διότι πρέπει να υπάρξουν κάποια όρια, κάποια όρια στο ωράριο εργασίας ε, του 7 και του 24ωρου. Δεν υπάρχει νομική βεβαιότητα εδώ, καμία νομική σαφήνεια. Ποιο είναι το ωράριο εργασίας Ποιες είναι οι ώρες, το ωράριο αναφοράς. Όλοι νομίζω ότι δίνουμε μια διαφορετική ερμηνεία. Επίσης αναφερθήκαμε στην, στο εύλογο χρονικό διάστημα κοινοποίηση. Αν θέλαμε σαφήνεια εδώ, θα έπρεπε την αρμοδιότητα αυτή να την αναλάβουν οι κοινωνικοί εταίροι. Και στα διάφορα κατάλληλα επίπεδα να γίνουν οι ανάλογες διαπραγματεύσεις. Όταν λέω για μας το θέμα των ε, ευάλωτων εργαζομένων είναι ζωτική σημασία. Το λέω γιατί στο άρθρο 9 η άκρος ευέλικτη εργασία θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον πιο καλοπληρωμένη. Δεν δίνονται κίνητρα στους ε, εργοδότες να χρησιμοποιήσουν αυτού του είδου τι συμβάσει. Γιατί λοιπόν να μην σκεφτούμε ένα ε, ορομίσθιο ε, ως για τις, για τις ή μετά το τρίμηνο να υπολογίζονται οι ε, ώρες που πραγματικά εργάστηκε κανείς στις εγγυημένες πραγματικές ώρες που περιλαμβάνει και η σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, εάν ε, κοινοποιηθεί κάτι σε έναν εργοζόμενο ε, και τον στείλουν σπίτι του ή τον στείλουν σπίτι του νωρίτερα, παρόλα αυτά πρέπει να πληρωθεί. Πρέπει να πληρωθεί για την ενημέρωση αυτή. Είτε εργάστηκε είτε όχι. Ένα άλλο θέμα είναι η μετάβαση σε ασφαλέστερη εργασία. Εδώ στο άρθρο 10 νομίζουμε το κείμενο δεν είναι αρκετά σαφές και ισχυρό. Για την ώρα έχουμε το θέμα του αιτήματο. Ένας εργαζόμενος μπορεί να αιτηθεί ό,τι θέλει από τον ε, εργοδότη του. Θα έπρεπε λοιπόν να μπορεί να ζητήσει να έχει ασφαλέστερη εργασία και ο εργοδότη μετά υποτίθεται ότι θα το εξετάσει και η άρνησή του μπορεί να βασίζεται μόνο σε αντικειμενικού λόγους που αφορούν την επιχείρηση. Αν δούμε όμω τα άρθρα για την επιβολή, άρθρα τα οποία τα βλέπουμε γενικώ θετικά, αλλά ένα σημαντικό θέμα Το θέμα είναι ε, η, νομική, καταγραφή. Ε, δηλαδή, να μην μπορούν τα κάτι να διαλέξουν από τα δύο παράλληλα συστήματα ότι τα βολεύει, γιατί μόνο η πραγματική ε, νομική καταγραφή θα βοηθήσει του εργαζομένου. Πάντως, σε κάθε περίπτωση το όλο κείμενο είναι ένα βήμα προοδού. Εάν προχωρήσει σωστά θα βοηθήσει του εργαζομένου να προστατευτούν και ελπίζουμε όλα αυτά να γίνουν στην δική σα θητεία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμεί Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Βαρνέκ. Και τώρα ο λόγος στον εισηγητή και στους σκιώδεις. Ο κύριος Καλβέτ Σαμπών πρώτος. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Μαρίτα και ευχαριστώ και τους ομιλητές. Νομίζω θα ήταν καλύτερα να ασχολούμαι με τον επιτύχο συμφωνία ειρήνης ε, μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράκ παρά να λύσω λιγάκι αυτά τα θέματα. Ε, μπας περιπτώσει. Δεν νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω σε όλα, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα θέματα τα οποία τράβηξαν την προσοχή μου και που είναι και θέματα κοινή ε, λογικής, ε, αφορούν και τις δύο πλευρές. Να αναφέρω κάποια παραδείγματα. Θέλω να υπογραμμίσω ότι δεν πρέπει να υπονομεύουμε την εφαρμογή των οδηγιών. Οι οδηγίες πρέπει να εφαρμόζονται. Βεβαίως υπάρχουν κάποια θέματα που θα πρέπει να είναι δεσμευτικά, όπως αναφέρθηκε και από την προλαλήσασα. Βεβαίως είπατε και πάρα πολλά άλλα. Εκείνο που θέλω να υπογραμμίσω είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή κατ' ουσίαν προσπαθούμε μέσα σε δύσκολες συνθήκες για τους Ευρωπαίους πολίτες προσπαθούμε να προσαρμόσουμε βασικά δικαιώματα για ενημέρωση στο βαθμό βέβαια που μπορεί να υπάρξει κάποια προβλεψιμότητα, να εφαρμόζουμε αυτό το δικαίωμα και να το προσφέρουμε σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Γιατί δεν είναι θέμα επικουρικότητας, είναι θέμα λογικής και ευφυούς αποκέντρωσης. Αυτό είναι το πρώτο, το πιο σημαντικό. Αλλά επίσης είναι αλήθεια ότι αυτά προχωράνε πολύ πιο πέρα από τον ορισμό του εργαζόμενου, που κατά την άποψή μου αυτό σημαίνει ανεξάρτητα με το τι θα κάνει κάθε κράτος για το κατά πόσον πρέπει να ληφθεί υπόψη ο εργαζόμενος, ο εποχικός ή μετά από αίτημα. Αυτό που είναι πολύ απλό, εάν υπάρχει εξάρτηση ανάμεσα στον εργαζόμενο και κάποιον που τον πληρώνει και του λέει κάνε αυτή τη δουλειά για μένα, αν υπάρχει αυτή η εξαρτησιακή σχέση, ο εργαζόμενος πρέπει να ξέρει τα βασικά θέματα για τη σχέση αυτή. Αν το δεχτούμε αυτό, νομίζω ότι μετά όλα τα άλλα μπορούν να προκύψουν στο, πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς στον κατάλογό μου έχω τον κύριο Ντένις Ράτκε, αλλά δεν τον βλέπω εδώ. Η κυρία Γιάσλοβεκ είναι παρούσα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Δεν ομιλώ εδώ εκ μέρους των άλλων, εκ μέρους άλλων, αλλά ομιλώ εξ ονόματός μου. Eh, Πρόεδρε, με μεγάλη προσοχή ακούσαμε τις τρεις παρεμβάσεις και ως σιώδης εισηγητής θέλω να υποβάλω παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Πρώτα-πρώτα Θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι πολύ καλή αφετηρία για να συζητήσει η Επιτροπή μας αυτή την πρόταση. Επίσης θεωρούμε ότι είναι πολύ θετική αυτή η πρωτοβουλία. Μπορεί να αποκτήσει έτσι ε, κάποιους ελάχιστους περιορισμούς για τα σχετικά δικαιώματα να τα θεσπίσει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τις νέες τάσεις που υπάρχουν. Πάντως πέραν αυτόν ερωτώ τι γίνεται με τον ε, ορισμό. Άκουσα τις επιφυλάξεις που υπάρχουν για το αν χρειάζεται ή όχι ευρωπαϊκός ορισμός. Αλλά πέραν αυτό το σχετικό με τον ορισμό που μας απασχολεί είναι το πεδίο εφαρμογής το βεληνικές αυτής της ε, οδηγίας. Η βεβαιότητα, η ασφάλεια που θα αφορά την εφαρμογή της ε, οδηγίας και για το κατά πόσον θα υπάρχουν δυνατότητες εφαρμογής αυτής της ε, οδηγίας. Ε, αυτό σίγουρα και έχει σχέση με τον ε, ορισμό. Αυτό που κάνει η Επιτροπή είναι να βαπτίζει η οδηγία την υπάρχουσα νομολογία. για να δούμε τι θα κάνουμε με τις μη αντιπροσωπευτικές μορφές συμβάσεων εργασίας και τι θα γίνει με τις συμβάσεις τις μηδενικέ, τι θα γίνει επίσης για την εργασία με πλατφόρμα να δούμε αν αυτό καλύπτει την πρόταση της Επιτροπής γιατί επιδέχεται η ρύθμιση και αυτή, αυτές, αυτές οι νέες μορφές εργασίας. Καλά, υπάρχουν κάποιε επιφυλάξει, αλλά νομίζουμε ότι τώρα μα προσφέρεται μια ευκαιρία να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να υπάρξει διαφάνεια στι εργασιακέ σχέσει. Madam McIntyre is e uh, δεν είναι εδώ από το ECR. Ούτε η κυρία Λόπες Μπερμέχο. Ούτε ο κύριος Τόμας Μέτσερη. Ούτε η κυρία Άτζια. Ζωέλ Μολέ. Ούτε εκείνη. Άρα, πάμε στην κυρία Γιάσο και πήγε το λόγο και κατόπιν θα πάρει το λόγο ο κύριος Μάνου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε σε μεγάλες λεπτομέρειες τη σκέψη των ειδικών όσον αφορά αυτό το σχέδιο οδηγίας να ευχαριστήσουμε επομένω τους ε, δύο εισηγητές για την ανάλυση ανά άρθρο. Μας αναφέρατε πώς θα εφαρμοστούν στην καθημερινή ζωή αυτές οι διατάξεις πάντως. Με εκπλήσει η στάση της Επιτροπής, της Κομισιόν γιατί υποτιμά τις ε, διαβλέψης των κοινωνικών εταίρων. Τον ρόλο τους στη χάραξη της κοινωνικής πολιτικής. Με τη σημερινή συγκυρία επιβάλλονται και θα γίνουν πολλές αλλαγές στην επόμενη πενταετία δεκαετία στην αγορά εργασίας, αγορά απασχόλησης, νέα μοντέλα, νέες μορφές απασχόλησης δεν έχει γίνει ολοκληρωμένη συζήτηση για αυτά. Οι νέες μορφές επιχειρήν. Για να δούμε πώς θα προετοιμαστούμε. Λέμε όλα τα ίδια και δεν προχωρούμε. Η κυρία Χάντβικ μας είπε για τις νέες μορφές εργασίας, για τις πλατφόρμες και Θέλω να ρωτήσω τους καλεσμένους μας. Ποιο είναι το κρίσιμο στοιχείο, πώς θα προετοιμάσουμε μια αξιόλογη ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις ε, νέες μορφές εργασιακών συμβάσεων. Μαν και μετά κύριος. Ο κύριος Μαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακριβώς όπως και η Ντανούτα και εγώ θα ήθελα να επισημάνω ότι κατά τη γνώμη μου, είναι μια καλή λύση να καλούμε τους εμπειρογνώμονες και βεβαίως όταν φέρνουν τόσες πολλές πληροφορίες μπορούμε και εμείς να μάθουμε πολλά πράγματα. Η Ντανούτα επισήμανε ότι είναι δύσκολο να μπορέσουμε να συνδυάσουμε όλες αυτές τις εμπειρίες μας. Εγώ θεωρώ στην Ευρώπη πρέπει να προσπαθούμε να επιτύχουμε προσέγγιση όσο γίνεται, αλλά να συμπεριλαμβάνουμε και τα κράτη-μέλη. Να μην έχουμε κανένα που να μπλοκάρει κάποια κατάσταση. Όταν όμως οι διαφορές είναι τόσο μεγάλες, τότε είναι λάθος λύση να λέμε ότι ξέρετε αυτό θα ρυθμιστεί στην Ευρωπαϊκή Οδό. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να συμπεριλάβουμε τους κοινωνικούς μας εταίρους, ακόμα και αν οι κοινωνικοί εταίροι δεν μπορούν να συμφωνήσουν, είναι σημαντικό να εκφραστούν. Αυτό δεν συμβαίνει σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Ε, και πολλές φορές ούτε κάνουμε τη δύναμη που υπάρχει και αυτό είναι λυπηρό. Εγώ θέλω να σας πω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να αποκτήσουν τη συνείδηση ότι η κοινωνική πολιτική είναι ένα αναπόσπαστο στοιχείο του κοινού ευρωπαϊκού, της κοινής ευρωπαϊκής πορείας. Άρα δηλαδή οφείλουμε να σκεφτούμε ε, το πώς μπορούμε να περιορίσουμε τις επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, πώς μπορούμε να επιτύχουμε να έχουμε συλλογικές συμβάσεις που θα συνάπτονται και πέρα από τα συνδικάτα. Γι' αυτό λοιπόν προβλέπονται αυτοί οι κανόνες. Τώρα, ε, οι διαφορές είναι μεγάλες, ε, πρέπει να συνεχίσουμε να συζητάμε όχι μόνο οι σκιώδεις, αλλά και εμείς όταν θα καταθέσουμε τις ε, τροπολογίες μας. τους χάρη παράγραφος 8 ε, για τις πολλαπλές ε, θέσεις απασχόλησης. Εκεί πρέπει να το δούμε λιγάκι. Στην παράγραφο υπερθυμών 10 υπάρχουν ε, διάφορες δυνατότητε. Αυτό που παίζει ρόλο εδώ είναι το predictable το προβλέψιμο. Να δούμε δηλαδή κατά πόσον είμαστε σε θέση να έχουμε ένα κανονισμό όπου θα αισθανόμαστε ότι εκεί μπορούμε να ανοίξουμε έναν ελάχιστο, έναν έστω μικρό διάβλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ε, τελειώνοντας θέλω να πω ότι η προστασία από την καταγγελία είναι κάτι πολύ σημαντικό Δεν μπορούμε να το αφήνουμε αρχαία κατά μέρος. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ε, στο βαθμό του δυνατού να έχουμε συλλογικές συμβάσεις, να μεριμνήσουμε, να το αισθανθούν αυτό οι πολίτες. Ε, είμαστε ένα κομμάτι αυτής της ε, παραγωγικής εξέλιξης, έτσι ώστε οι άνθρωποι να πληρώνονται πραγματικά καλά ε, και στο τέλος να υπάρχει και να επικρατήσει δικαιοσύνη και να μην καταλήγουμε μόνο σε πανηγυρικούς. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαν. Η κυρία Ευχαριστώ πολύ τους εμπειρογνώμονες που ήρθαν εδώ. Ε, κρίμα που δεν μπόρεσαν να έρθουν οι άλλοι δύο, αλλά με πάση περιπτώσει σας ευχαριστώ πολύ για αυτά που μας είπατε. Εγώ μπερδεύτηκα λίγο. Ίσως λοιπόν μπορείτε να με βοηθήσετε να τα ξεμπερδέψω. Όσον αφορά τον ορισμό του εργαζόμενου. Διότι... Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι δικηγόρος. Ίσως λοιπόν αυτό να εξηγεί και γιατί κάνω αυτή την ερώτηση. Η Κομισιόν καθιστά απόλυτα σαφάς, σαφές ότι το μόνο που κάνει στον ε, ε, ορισμό του εργαζόμενου είναι ότι εφαρμόζει την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και διαρωτώ με, πώς είναι δυνατόν να τα γεφυρώσετε αυτά με το αυστριακό εργατικό δίκαιο. Γιατί η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και αυτή θα οδηγεί σε συνέπειες, συγκεκριμένες συνέπειες στα κράτη-μέλη. Αυτό λοιπόν είναι ο γρίφος που με προβληματίζει. Αυτό κάνει η Κομισιόν, απλά δηλαδή εφαρμόζει την νομολογία και αν δεν το κάνει αυτό τότε πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφύγει να δημιουργούνται προβλήματα όπως παραδείγματος χάρη αυτά με το αυστριακό δίκαιο. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και κάτι άλλο. Οι κοινωνικοί εταίροι εκτιμούν όλες αυτές τις συζητήσεις ε, που οδηγούν ε, ε, σε συμφωνίες κοινωνικών εταίρων. Γιατί πρέπει να σας πω ότι καμία από τις οδηγίες που επιτεύχθηκαν, όπως αυτή για την κομμωτική, δεν μεταφράστηκε ε, σε ευρωπαϊκή νομοθεσία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διερωτώ με αν τελικά είχατε χρόνο για να σωστό κοινωνικό διάλογο. Και αυτή την ερώτηση την εκφράζω στον εκπροσώπο, εκπρόσωπο του Business Europe. Αν είχατε λοιπόν χρόνο, αυτό πώς θα επηρέαζε το περιεχόμενο και οι εργαζόμενοι με επισφαλείς ε, συμβάσεις πώς θα μπορούσαν να επωφεληθούν. Επίσης, ε, θα ήσασταν πρόθυμοι να βάλετε στο τραπέζι όλες σας τα χαρτιά. Ο εκπρόσωπος των Ευρωπαϊκών ε, Συνδικάτων ε, θα μπορούσε να μας πει κατά πόσον αυτό θα ήταν ικανοποιητικό ή όχι. Γιατί τώρα Απλά ακούμε, ακούσαμε λίγο ότι ενδεχομένως θα ήταν δυνατόν. Τι θα ήταν αυτό που θα ήταν ίσως δυνατόν και τι θα άλλαζε τελικά στη ζωή των απλών ανθρώπων στην Ευρώπη. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Και τώρα να ξαναπάμε στους... Α, όχι. Προηγουμένως ο λόγος στον κύριο Μπάουνλε που είναι εισηγητή στην ΕΟΚΕ. Και μετά θα πάμε στους εμπειρογνώμονες. Γιατί έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις να σας κάνω. Κύριε Μπάουνλε. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσω. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τους τελευταίους μήνες είχαμε συζητήσεις ανάμεσα στους εργοδότες και τους εργαζόμενους στην δική μας την Επιτροπή που έμοιαζαν πράγματι πάρα πολύ με ειρνευτικές διαπραγματεύσεις. Τελικά βέβαια καταλήξαμε σε ένα συμβαστικό κείμενο και πολύ ευχαρίστως να σας ενημερώσω. Πέρασε αυτό το κείμενο από τα τμήματα και την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια θα ληφθεί η τελική απόφαση. Και η γραμμή που ακολουθούμε είναι περίπου αυτή που είπε ο κύριο Τόμας Μαν. Εμείς θα θέλαμε το θέμα αυτό να λυθεί με διαπραγματεύσεις μέσα από τους κοινωνικούς εταίρους, ε, σε εθνικό επίπεδο βέβαια, αλλά εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό παντού στην Ευρώπη, γι' αυτό και στηρίζουμε την νομοθετική πράξη της Επιτροπής και την πρόταση. Κατά τα άλλα, θέλω να αναφέρω ότι όσον αφορά τον ορισμό του εργαζόμενου έχουμε κάποιες επιφυλάξεις κατά πόσο μπορεί αυτός ο ορισμός να ισχύει και για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες. Εμείς πιστεύουμε ότι ο αλγόριθμος ε, μπορεί να επηρεάσει ε, τη ζωή ενός ανθρώπου ακριβώς όπως και οι γραπτές ή προφορικές ε, οδηγίες. Γι' αυτό λοιπόν οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες που δεν είναι ακριβώς ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. Τον ορισμό του εργοδότη και εκεί πρέπει να υπάρξει μία διευκρίνηση ως προς την υποχρέωση ενημέρωσης θεωρούμε ότι την εποχή της ψηφιοποίησης ε, θα πρέπει κανείς να είναι ενημερωμένος από την πρώτη μέρα ε, για τις συνθήκες της σύμβασής του όταν ξεκινάει η εργασία του. Αν δεν είναι πρέπει να δούμε γιατί δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Πάντως πιστεύουμε ότι σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να επικρατεί ευελιξία και θέλουμε να επισημάνουμε ότι όταν ανακοινώνονται οι συλλογικές ε, συμβάσεις ε, κατ' ουσίαν ε, θα πρέπει να προκύπτουν και εφαρμόσιμες λύσεις που δεν επιβαρύνουν τον εργοδότη. Όσον αφορά τώρα τις συνθήκες εργασίας, εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν συμβάσεις μηδενικών ορών ε, στη Γερμανία μου έκανε τεράστια εντύπωση. Είναι δυνατόν να συναυθούν τέτοιες συμβάσεις. Τώρα όμως ευτυχώς ε, το θέμα λύθηκε, συζητήθηκε στις ε, διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης και αποφασίστηκε ότι θα λυθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι σε αυτές τις μορφές απασχόλησης είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι. Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε εργασία ε, και ε, απασχολούνται για πάνω από 6 μήνες έχουν δικαίωμα ενημέρωσης και έχουν και δικαίωμα για να περάσουν σε ασφαλή απασχόληση εφόσον βέβαια αυτή υπάρχει στην εταιρεία. Και τελειώνοντας θέλω να σας πω ότι για μας ε, είναι πολύ σημαντικό αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καταρχήν τη θεωρούμε σωστή η πρόταση αυτή να συζητηθεί σε εθνικό επίπεδο από τους κοινωνικού εταίρους και εκείνοι να καταλήξουν στις τελικές ρυθμίσεις. Αυτό κατά την άποψή μας είναι ο καλύτερος δρόμος. Ευχαριστώ. Λόγο για να απαντήσει σε κάποια από τα θέματα που ε, ανέκυψαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους εμπειρογνώμονες και όλα τα μέλη. Να θυμίσω ίσως ότι όπως αναφέρθηκε η πρόταση αυτή <coughs> είναι το όντι η συνέχεια που δόθηκε στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων που εγκρίθηκε πέρσι τον Νοέμβριο και επισήμω ε, έγινε διάγγελμα για αυτόν στον Κέτεμπορκ τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ε, μιλάμε για εξισορρόπηση του επαγγελματικού με τον προσωπικό βίο και την πρόταση της Επιτροπής για Σύσταση στην πρόσβαση, για την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για όλους. και προκειμένου να υπάρχει επαρκή κοινωνική κάλυψη για τους αυτοαπασχολουμένους. Όπως ε, σημειώθηκε, πρόκειται για μια σημαντική απόκριση για την αύξηση της, ε, στην αύξηση της παράτυπης εργασίας. Τα τελευταία δέκα χρόνια οι μισές από τις νέες θέσεις εργασίας ήταν άτυπες. πολύ σύντομη, μερικής, ε, μερικού χρόνου εργασίας, πολύ σύντομης διάρκεια συμβάσεις, ε, λίγο πολύ η επισφάλεια επιτάθηκε. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπή είναι να βρει ένα σημείο ισορροπίας μεταξύ της απαραίτητη ευελιξίας στην αγορά εργασίας και την ε, απαραίτητη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω των νέων μορφών Προστατεύοντα βεβαίω και τους ευάλωτου ε, και όσου βρίσκονται σε επισφαλείς θέσεις. Αυτό μας φέρνει στο θέμα του πεδίου ε, και του ορισμού του εργαζομένου που προστατεύεται. Ένα από τα βασικά ε, ζητήματα που προέκυψαν. Μια από τις βασικές μορφές επισφάλειας είναι να μην έχει κανείς το καθεστώς του εργαζομένου. Καν αυτό το χαρακτηρισμό και το εντόπισαν πολλοί από τους ομιλητές μας. Αυτό που πρότεινε εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να κωδικοποιήσει κάπως μία ε, ευρωπαϊκή έννοια ε, που έχει ουσιαστικά επικρατήσει και την έχει διατυπώσει το δικαστήριο στην ομολογία του από το 1996 σε πολλές αποφάσεις, καλύπτοντας πολλές αποφάσεις για την κοινωνική προστασία έκτοτε. Ιδίω για να οριστεί εάν ένας οικονομικός ενεργά ε, πολίτης είναι ασχέτως του καθεστώτος του αυτοπροσχαλουμένου μισθωτού εργαζόμενος ή όχι. Αυτή η διατύπωση συνάδει. <coughs> συνάδει Ε, με, την επίσημη, ε, με τον επίσημο ορισμό για τον εργαζόμενο. Όμως αυτό που σημαίνει αυτό είναι ότι το προσωπικό πεδίο του, της οδηγίας θα πρέπει να μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία και εκεί να οριστεί τι είναι ο εργαζόμενος. Εάν η εθνική νομοθεσία δεν καλύπτει όλες τις ε, μορφές θα ισχύει και θα υπερισχύει ο ορισμός της οδηγίας. Οι εγχώροι εργαζόμενοι λοιπόν εφόσον εργάζονται ε, σε πλατφόρμες αυτό μπορεί να επιληθεί στις περαιτέρω ρυθμίσεις για τη μεταφορά της οδηγίας. Αυτό που υποκρύπτει αυτή η λογική είναι ότι ακριβώς θα έχουμε μια οδηγία που θα αντέξει στο μέλλον για να καλύψει νέες μορφές εργασίας που ακόμη δεν έχουν αναπτυχθεί. Γι' αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε να πούμε ότι η οδηγία αυτή είναι οδηγή. Γι' αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε να πούμε ότι η οδηγία αυτή είναι οδηγία που θέλει να προστατεύσει την εργασία σε πλατφόρμες. Θέλει να προστατεύσει όλες τις μορφές εργασίας και όποιον εμπίπτει στον ορισμό του εργαζομένου. Ε, οδηγία θέλει να προστατεύσει την εργασία σε πλατφόρμες. Θέλει να προστατεύσει όλες τις μορφές εργασίας και όποιον εμπίπτει στον ορισμό του εργαζομένου. Ε, το ρόλο των κοινωνικών εταίρων και λυπούμεθα που δεν ήταν δυνατό σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι δύο βασικοί ευρωπαϊκοί εταίροι να ε, περάσουν σε διαπραγματεύσει ε, για την εκπόνηση τη πρόταση. Η πρόταση όμω έλαβε υπόψη όλε τι ε, προθεσμίε που προβλέπει η συνθήκη. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ουσία, πολύ βασική, και σίγουρα έπρεπε να υπάρχει κατάλληλη διαπραγματευτική βάση εντό των προθεσμιών που προβλέπει η συνθήκη. Όμω, οι λόγοι που υποβάλλουμε αυτή την πρόταση ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι όντω αντιμετωπίζει του ευπαθεί εργαζομένου και τι δυσκολίε τη αγορά εργασία που γίνονται όλο ένα και πιο έντονε. Και θα τα βάλουν στο νομικό του σύστημα. μπορούν να τα μεταφέρουν με τρόπο που να προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία. Λόγω χάρη διατύπωση ή απλοκο χρονικό διάστημα σημαίνει συγκεκριμένα ότι αυτή την έννοια μπορούν να την ερμηνεύσουν ανάλογα με μια ε, σειρά από δικαιώματα με τρόπο διτό. Πρώτον, ε, τους εργαζομένους όπως αδρά ορίζονται, δεν είναι το δικαίωμα να ενημερωθούν για τα βασικά στοιχεία της εργασιακής τους σχέσης, ε, είναι ε, των πραγμάτων δίκαιο να γνωρίζει κανείς ξεκινά να ενημερωθούν για τα βασικά στοιχεία της εργασιακής του σχέσης ε, είναι των πραγμάτων δίκαιο να γνωρίζει κανείς ξεκινά και στο τρίτο κεφάλαιο της πρότασης υπάρχει ένα σύνολο από βασικά ουσιαστικά δικαιώματα είναι ένα θέμα αυτό που χρήζει περαιτέρω εξέτασης, όμως είναι σημαντικό να διαθετηθεί. Σκεφτήκαμε λοιπόν εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, ώστε να συμφωνήσουν διαφορετικό σύνολο δικαιωμάτων εφόσον το επιθυμούν, εκεί όπου οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται. Να είναι ένας πολλαπλός εργοδότης. Η τάση όμως αυτή διαφαίνεται ήδη σε πολλές εργασιακές σχέσεις ε, με τα πάνω από έναν φορέα που που έχει την ε, ιδιότητα του εργοδότη, αλλά αυτό εναπόκειται στα κάτι μελη Επίση είναι να θεσπίσει και να εδραιώσει δικαιώματα για όλου του εργαζόμενου. Το άρθρο 17 υπάρχει ένα τρόπο προάσπιση που προβλέπεται για τα δικαιώματα αυτά, εφόσον απειτέω σχόλιο στην οδηγία για την ε, εργασία. Ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει ο εργοδότης να απαντά γραπτός σε αίτημα ε, του εργαζομένου για πιο προβλέψιμη, ασφαλέστερη θέση εργασία. Δεν εξισορρόπηση επαγγελματικού και προσωπικού βίου. Σε κάθε περίπτωση καλωσορίζουμε όλα σας τα σχόλια. Θα τα μελετήσουμε προσεκτικά. Θέλουμε να συνεργαστούμε αυτή τη και αν υπομονούμε να συνεργαστούμε με την Επιτροπή σας για να επιτύχουμε ψηλό επίπεδο προστασίας για όλους τους Ευρωπαίους εργαζομένους. Ευρωπαϊκό Εργατικό δίκτυο Μας για να δούμε τι έχουν να απαντήσουν. Όποιος θέλει εξημών μπορεί να ξεκινήσει. ευχαριστώ. Και φυσικά το κάνει. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη τις εξής δύο αποφάσεις. Η πρώτη είναι του 86. Πρώτη απόφαση σε σχέση με την ελευθερία διακίνηση εργαζομένων κυκλοφορία τους που είναι βέβαια κάτι διαφορετικό. Μιλούμε εδώ για ενοχικό δίκαιο, δεν μιλούμε για την ελεύθερη κυκλοφορία. Στη δεύτερη απόφαση έχουμε την σχέση μεταξύ μιας καλόγριας και του τάγματος στο οποίο ανήκε. Ε, δεν νομίζω ότι αυτό είναι και πολύ σχετικό με τα όσα συζητούμε. Ε, άρα πώς αυτά να αποτελούν την αφετηρία ούτως ώστε να πάμε για έναν ορισμό εκατοντάδες δικαστικών αποφάσεων σε σχέση με το θέμα του ορισμού. Οπότε στις χώρες μας ξέρουμε τι γίνεται με τους δημοσιογράφους, τι γίνεται με τους διαφημιστές, ε, τους ασφαλιστές, τι γίνεται επίσης ε, με τους χαρακτηριστικά αυτών των ε, ε, αυτοαπασχολουμένων και άρα τώρα πάμε για ένα νέο ορισμό, αλλά προσοχή να μην πέσουμε σε έλλειψη ασφαλείας δικαίου και θολούρα όσον αφορά την εφαρμογή του ορισμού στις χώρες. Κεντρώνουμε την προσοχή μας στο πώς θα ενημερώνονται οι πληροφορίες οι οποίες ε, δίνονται στον ε, εργαζόμενο. Πολλά είναι τα σχετικά παραδείγματα. Να είναι η κατάσταση νομική ξεκάθαρη, όχι ασαφής όπως την πρόταση της Κομισιόν να δούμε τι γίνεται με τους οργανισμούς, στις πλατφόρμες και όλα αυτά θέλουμε να προετοιμαστούμε. Και θα πρέπει να σας πω και να τονίσω ότι μας εξέπληξε η πρόταση της Κομισιόν. Θα λείπει, όπως είπα επανειλημμένα, των υψηλών δεξιοτήτων και υψηλέ αμοιβή εργαζομένων. Και η συνάδελφο τι γίνεται με που χτίζονται από το ευάλωτο, αλλά η ίδια δουλειά σε κάποιες χώρες δεν επιβάλλεται, είναι ελεύθερη επιλογή, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο σε τη εργασία. Και υπάρχουν, ασάφιος τα λέει εδώ πέρα. Αλλαγή από μερική απασχόληση μέχρι πλήρη απασχόληση μπορεί να, προσθέσει ώρες. Υπάρχει πλήρη ρύθμιση, στεγανή ρύθμιση. Θέλει να αλλάξει το καθεστώ η, Κομισιόν. Ε, ας μας ρωτήσει πρώτα, να μα ρωτήσει να δει αν Είπατε μάλλον ότι είχαμε νέα μήνες να κάνουμε τη διαβούλευση. Ε, όχι. Μας δώσατε ένα μήνα. Αυτό είναι αδύνατο για εμάς τους κοινωνικού εταίρους. Για να δούμε τώρα όσον αφορά τον ορισμό. Χαβιέρ Λόπες, είστε ακόμα εδώ. Μάλιστα. Γεια σας, γεια σα. Γιατί υπάρχει εδώ πέρα κάποια διάκριση ότι θα πρέπει να είναι εθνικές αρμοδιότητες και από τη δική μου χώρα, από την Δανία, η κοινωνική εταίρεια, κάνω κάποια συμφωνία δοκιμαστική, πλατφόρμα. να δούμε ποιοι είναι αυτοαποσχολούμενοι, ποιοι δουλεύουν για την πλατφόρμα. Αν στην πράξη τη ισχύει και δεν θα πρέπει να έχουμε μόνο διάστατη κοινωνική νομοθεσία, να δανειζόμαστε στοιχεία από άλλε οδηγίε, γιατί έτσι παγώνει μια κατάσταση. Γίνεται άκαμπτη δεν μπορούμε έτσι να προσαρμοστούμε στη μορφή που θα τα πράγματα στο μέλλον επίσης. Τι να δω τον Γίνεται άκαμπτη. Δεν μπορούμε έτσι να προσαρμοστούμε στη μορφή που θα τα πράγματα στο μέλλον επίσης. Τι να το των κρατών μελών. Μπορεί να υπάρχει κάποια παρέκκληση για κάποιους ευκαιριακά εργαζομένους. Άλλο θέμα αυτό. Εμείς θα προτιμούσαμε για την έκθεση Refit που διαπιστώνει προβλήματα, θα θέλαμε λέγω η Κομισιόν να πάει στα κάτι με υπάρχουν προβλήματα και να ζητήσει να προβούν σε προσαρμογή. Υπάρχουν νέες μορφές ευκαιρικής εργασίας, άρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εξασφαλίσουμε το ότι δεν θα έπρεπε να είμαστε υπερβολικά άκαμπτοι και από τα μεριά όμως, να καλύψουμε αυτές τις μορφές εργασίας εκεί που είναι λογικό. Να γίνει ευρωπαϊκή ρύθμιση. Όμως, να μην βιαστεί κανείς να τα βάλει όλα αυτά σε μια οδηγία, γιατί άμα το κάνει αυτό, μετά ό,τι γίνεται δεν ξεγίνεται. Τα σε ευχαριστούμε. Οδηγίας. Θα πρέπει να καλυφθεί και αυτό από την οδηγία, επομένως έχει το σημασία το άρθρο 8. Δεν μπορεί ο εργοδότης να μπορέσει την παράλληλη απασχόληση. Και αντίστα προς το ζει. Για να τα βγάλει κανείς πέρα χρειάζεται δυστυχώς περισσότερες συμβάσεις εργασίας. Ώστε να καλύψουμε και την δυνατότητα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων σε διαφορετικά επίπεδα, ό,τι σημαίνει αυτούς τους τύπους μορφότυπους τέλο πάντων. Να πρέπει να δούμε σε τι μορφή θα πρέπει να συνέρχονται. Και βέβαια αυτός ο τύπος των διαπραγματεύσεων και επαφών θα ήταν χρήσιμο εργοδότες οι οποίοι έχουν υποχρεώσεις και δικαιώματα Και... Τώρα το τι επιδέχεται διαπραγματεύσει. Υπάρχει η ρύθμιση της μετάβασης από το ένα είδος στο άλλο. Αλλά θα πρέπει ο εργοδότης να το φροντίσει αυτό. Άρα με την οδηγία σε δεν μπορεί κάποιος να έχει σύμβαση για δεκάωρη και αν θέλει να πάει σε κάποια που ε, Να υποβάλουν ερωτήσεις. Νομίζω ο Ενρίκε έχει ζητήσει το λόγο. Να υποβάλουν ερωτήσεις. Νομίζω ο Ενρίκε έχει ζητήσει το λόγο. Αλλά επίσης έχουμε εδώ και τον Ισπανό σκιώδη ε, εισηγητή που είναι ο μόνος που παρίσταται εδώ να σας τα πω στα ισπανικά. Μια που η Επιτροπή μας δεν είναι Επιτροπή για διαπραγματεύσεις και εγώ είμαι εισηγητή